Ζητήθηκε να <clears throat> προστατευτεί αυτή η ασυλία, όπως θα σας είναι γνωστό. Uh, και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια, στην ημερήσια διάταξη. Και σύμφωνα με, με το άρθρο 4, εδάφιο 1 και εδάφιο 4, σημειώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την κατάσταση πραγμάτων και με βάση το άρθρο 3 εδάφιο 2 η κυρία Μόνικα Κλέφερ Πρέντεγκαστ και Σάντο Τέβο θα είναι τα νέα μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέχρι την επαλήθευση των, της διαπίστευσής τους και με την υπογραφή μιας γραπτής δήλωσης ότι δεν έχουν άλλο αξίωμα σύμβατο με το αξίωμα του Ευρωβουλευτού θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες με πλήρη δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αρμόδιες αρχές της Σλοβενίας με ενημέρωσαν ότι ο κ. Ζόραν Τάλερ αντικαθίσταται από Κλέφερ από την ε, από τον Απρίλιο ήδη και οι Ιρλανδικές αρχές ανέφεραν ότι ο κύριο Κέλλη αντικαθίσταται από τον κύριο Φιλ Πρέντεγκάστα και μάλιστα από την 13η Απριλίου 2011. Οι αρμόδιες φινλανδικές αρχές είπαν ότι η Δημοσύνη εξελέγει στο Φινλανδικό Κοινοβούλιο και έτσι πάβει να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 26η Απριλίου 2011. Θα αντικατασταθεί από την 26η Απριλίου 2011 από τον κύριο Σαμκο Πέρχο. Διερωτώ με αν τα νέα μέλη βρίσκονται στην αίθουσα. Ίσως θα μπορούσαν έτσι να αυτοπαρουσιαστούν. Παρακαλώ. Well, thank you very much. The next. Thank you very much. And the third colleague. Third colleague. Και ο τρίτος συνάδελφος. Παρακαλώ. Δεν βλέπω να παρίσταται. Εντάξει. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Και σύμφωνα με το άρθρο 3, εδάφια 3 και 4, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων